Benissimo, Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Ζητώ συγγνώμη για την ε, αργοπορία, αλλά είχε πάρα πολύ πάρα πολύ ε, ε, κίνηση στις Βρυξέλλες. Ξέρετε, περνάνε τα σκουπιδιάρικα πρωί και γίνεται χαμός. Σταματάνε τα πάντα. Λοιπόν, καλημέρα. Ε, καλώς ορίσατε σε αυτήν την συνεδρίαση στην οποία προεδρεύω στη θέση του Προέδρου Ταγιάννη ε, έχουμε διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά τα οποία μπορείτε να ακούσετε και να μιλήσετε ε, σχέδιο ημερησία διατάξεως, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, να εγκριθεί. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασής μας ε, θα εγκριθούν τα πρακτικά αύριο στις 10, εκτός και εάν υποβάλλεται εντωμεταξύ στη γραμματεία κάποιες ε, τροποποιήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνεδρίαση η οποία είναι έκτακτη, αποφασίστηκε στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας πρώτα απ' όλα. Ε, σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητήσουμε για τη μεταρρύθμιση ε, της ε, Τη συνέλευσή μα στην. Ε, θα ασχοληθούμε βέβαια και με το τι θα γίνει στην ε, Ρώμη την επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά την Ολομέλεια της Ρώμης, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουμε επανειλημμένα συζητήσει, κυρίως δε στην τελευταία μας συνάντηση. Κυρίως να μην λησμονούμε ότι πέρα από τη μεταρρύθμιση της συνελεύσεως, η Ολομέλεια ε, θα εγκρίνει και τις ετήσιες συστάσεις της Επιτροπής καθώς επίσης και θα ορίσει και τη νέα Προεδρία ε, Βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν Κοινοβούλιο είναι κυρίω ε, κυρίως να εγκρίνουμε τις συστάσεις του συναδέλφου Ρενάτο Σόρου όσον αφορά ε, την πορεία της Ευρώπης σε σχέση με τη Μεσόγειο. Αυτή η σύσταση κατά την άποψή μας είναι σημαντική έτσι ώστε να ενισχυθεί ε, ο δημοκρατικός έλεγχος της Ένωσης για τη Μεσόγειο και έτσι ώστε να ολοκληρωθούν ε, τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να διασφαλιστεί και η πρόοδος αλλά ε, και η διαφάνεια όλων των βημάτων. Ε, έχουμε υποβάλει κείμενο, έχουν υποβληθεί τροπολογίες, ελπίζω να φτάσουμε στη Ρώμη με ένα αποδεκτό συμβιβαστικό κείμενο. Όσον αφορά την επόμενη συνεδρία θα γίνει στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, στην άλλη όχθη δηλαδή, βάση και της αρχής της εναλλαγής Βορρά-Νότου που εφαρμόζεται εις την Προεδρία της Συνέλευσης ε, της Ένωσης για την Μεσόγειο εγώ δεν θέλω να πω αν μου αρέσει περισσότερο ε, ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος ή μία ή η άλλη υποψηφιότητα αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε για το θέμα αυτό σήμερα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος Ταγιάννη ε, ίσως κληθεί να επιλέξει ανάμεσα από τις δύο χώρες. Τέλος, διάσκεψη των προέδρων. Ξεκίνησε, εγγενιάστηκε το 2013 στη Μασαλία όπως ξέρετε ε, υπό την αιγίδα και προεδρία του, ε, του ε, Προέδρου Μάρτιν Σούλτς. Ελπίζω ότι από την διάσκεψη κορυφής η οποία θα έχει αυτή τη φορά ε, σαν θέμα την ανεργία και την ε, μετανάστευση να εξαχθούν ε, σημαντικά συμπεράσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε παρατηρήσεις επί των σημείων αυτών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τις υποβάλλετε άμεσα. Τώρα δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο κεντρικό σημείο της ε, σημερινής μας ε, συνεδρίασης που είναι η μεταρρύθμιση της συνελεύσεως υπό την όθηση της συναδέλφου Τιτσιάνα Μπεγκίνη, η οποία είναι πρόεδρος ε, της ε, ομάδας ε, που ασχολείται με το καταστατικό και τα οικονομικά ε, της συνελεύσεως ξεκινήσαμε ήδη από πέρσι μία συζήτηση όσον αφορά τα διάφορα θέματα της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως την συνάδελφο Μπεγκίν για την μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει τους τελευταίους μήνες. Η κυρία Μπεγκίν θα μας δώσει πληροφορίες τώρα σχετικά με την πορεία των εργασιών οι προτάσεις αυτές ε, λόγω της αντίθεσης κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Ένωσης Μεσόγειο κυρίως όσον αφορά ας πούμε την ε, μείωση του αριθμού των επιτροπών επίσης της αλλαγής της αρχής της υποχώρησης κτλ. δεν έχουν οι παρατηρήσεις αυτές γίνει αποδεκτές όλες. Εν πάση περιπτώσει αποτελούν σημείο εκκίνησης της συζητήσεως και βεβαίως ε, θα ληφθούν υπόψη τέσσερις κεντρικοί στόχοι. Πρώτον, πλήρη συμμετοχή στη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης για τη Μεσόγειο και στην ευρωμεσογειακή πολιτική. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να τοποθετηθεί ε, η κοινοβουλευτική συνέλευση ως κεντρικό σημείο κοινοβουλευτικής αναφοράς ε, που θα ασχοληθεί με σημαντικά θεμελιώδη ζητήματα για το μέλλον της ενώσεως όπως ας πούμε το θέμα των μεσογείων, των ε, προσφύγων, επίσης ε, βιώσιμες εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και κλιματικές αλλαγές. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να ασκήσει έναν ρόλο δημοκρατικού ελέγχου, πρωτοβουλίας και προτάσεων όσον αφορά στους στόχους της Ένωσης για τη Μεσόγειο τέταρτο και τελευταίο θα πρέπει να επιτρέψει στην ανανεωμένη κοινοβουλευτική συνέλευση να συμβάλλει αποτελεσματικά στις κοινέ προσπάθειες σταθερότητας και βιώσιμης δημοκρατικής ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην λησμονούμε αυτά τα τέσσερα σημεία όταν θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το μέλλον της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπεγκίν για να δούμε μέχρι πού έχουμε φτάσει όσον αφορά τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους κοινοβουλευτικούς μέλου της ε, ε, συνελεύσεως από τον Μάρτιο και μετά. Με τον τρόπο αυτό και μέσω της συζητήσεως θα προσπαθήσουμε προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους κοινού τόπους έτσι ώστε να φτάσουμε καλά προετοιμασμένοι ε, στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπεγκίνη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να ασχοληθώ, να σας αναφερθώ στις ε, ε, ε, συζητήσεις που έχουμε κάνει και τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ε, στην ουσία συζητούμε τώρα για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από μακρά προπαρασκευαστική εργασία. Στο, σε, σε παράρτημα σας έχω ήδη δώσει όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εργασίες που έχουν λάβει χώρα. Έχουν προκύψει και κάποιες τροποποιήσεις βάσει της συζήτησης της 30 Ιανουαρίου αλλά και του μηνός Μαρτίου. Οι προτάσεις οι οποίες υπευλήθησαν λάμβαναν υπόψη ε, την συνένεση των ε, ε, μελών όσον αφορά τέσσερα σημεία. Τον αριθμό των πέντε που δεν θα πρέπει να αλλάξει, η αρχή της υποχώρησης που δεν θα πρέπει, παραχώρησης που δεν θα πρέπει να αλλάξει, επίσης τα άρθρα 14 και 15 που δεν θα πρέπει να αλλάξουν και τέλος η συνεισφορά ε, στο προϋπολογισμό που θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική καθώς επίσης και το σύστημα των κυρώσεων βάσει του άρθρου 14 για όσους ε, δεν ε, καλύπτουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησαν στέλνοντας προτάσεις τροποποίησης έγκαιρα εκτός από την Πολωνία η οποία έστειλε παρατηρήσεις οι προτάσεις οι οποίες βρίσκονται στο φάκελό σας ε, έχουν 73 τροπολογίες. Οι τροπολογίες ε, αυτές μπορώ να, να σας τις παρουσιάσω συνοπτικά ως εξής. Όσον αφορά τον κανονισμό της ε, συνέλευσης υπογραμμίζω ότι ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μονάχα το Λαϊκό Κόμμα έχει στείλει προτάσεις τροποποίησης. Οι άλλες τρεις αντιπροσωπείες έστειλαν μεν τροπολογίες αλλά δεν μας επιτρέπουν να βρούμε κάποια κοινά θέματα όσον αφορά τις συνεισφορές στη Γραμματεία και τις ε, κυρώσεις. Η αντιπροσωπεία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή του Λαϊκού Κόμματος, ε, ζήτησε μέσω του άρθρου 4, παράγραφος 5α, σελίδα 3 του εγγράφου, να δώσει λοιπόν αρμοδιότητες στις Επιτρόπου από αποστολές. Άρθρο 4, εδάφιο 6, σελίδα 4. Όσον αφορά τώρα τις μεταφορές αρμοδιοτήτων βάσει του άρθρου 5 σελίδα 4 του εγγράφου η Πολωνία δεν δέχεται αυτήν την μεταβίβαση. Όσον αφορά τώρα τις εκκυρώσεις για αυτούς που δεν καλύπτουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις υπευλήθη η πρόταση να μην ε, κρατήσει ε, αυτός ο οποίος δεν έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του ε, την θέση του. Η Ιταλία όμως δεν συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί με τη θέση του Λαϊκού Κόμματος. Η Ιταλία θεωρεί ότι μπορούν να αντικατασταθούν βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 7, ε, σελίδα 7 του εγγράφου σας ε, να αντικατασταθούν λοιπόν από τους επιτόπου υπαλλήλους. Τέλος, όσον αφορά τη σύνθεση της γραμματείας. Η Ιταλία και η Γερμανία δεν συμφωνούν με την προτινόμενη απλούστευση. Η Ιταλία θέλει ε, η γραμματεία να έχει έναν γενικό γραμματέα και έναν λογιστή. Η Γερμανία δεν θέλει να τροποποιήσει το άρθρο 15 υφιστάμενο σελίδες 7 και 8. Η Ιταλία λέει τουλάχιστον για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει οπωσδήποτε την θέση του λογιστού βάσει του άρθρου 17 σελίδα 8 του εγγράφου να καλύπτεται από υπάλληλο του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επ' αυτού να έχω την άποψή σας, όπως φυσικά και όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ε, ιδιαίτερα ενεργή ε, στην διάρκεια της συνέλευσης ε, και μάλιστα πήρε τόσο μεγάλη θέση που τα τελευταία χρόνια τα υπόλοιπα κοινοβούλια δεν έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργητικότητα. Όσον αφορά τον οικονομικό κανονισμό, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Οι τροπολογίες που έχουμε λάβει δεν βασίζονται στα τέσσερα άρθρα του νέου ε, ε, ε, κανονισμού, αλλά ε, πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες πολύ ε, ε, απομακρύνονται από την αρχική μας θέση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στη Ρώμη να γίνει συζήτηση, διότι κάθε μία πρόταση είναι πάρα πολύ καλή και ενδιαφέρουσα, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ απλό να βρούμε κοινό τόπο, κυρίως όσον αφορά τον γενικό κανονισμό όσον αφορά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και στόχος της σημερινή ε, συζήτησης, γιατί θα πρέπει να συντονιστούμε επ' αυτού, πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ε, ε, ε, δεν βρίσκουν συμφωνία ανάμεσα στις ε, προτάσεις ε, του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών. Το πρώτο είναι η πρόταση του, για το σχέδιο του προϋπολογισμού που πρέπει να υποβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίε για τους σοσιαλιστές και για, τους, για το ΕΛΚ. Το ίδιο και η αρχή ρύθμισης του προϋπολογισμού. Μόνο το ΕΛΚ όμως λέει τι θα γίνει όταν η Ολομέλεια μέλη λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση ε, του οικονομικού έτους. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, η πρόταση του ΕΛΚ ε, διατηρεί το άρθρο 5, δηλαδή διαβούλευση ε, με, το, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, όσον αφορά το σχέδιο του προϋπολογισμού, όχι ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όσον αφορά το διαβριμένο Προεδρείο, το ΕΛΚ λέει ότι το διαβριμένο Προεδρείο θα πρέπει να εγκρίνει ε, τον προπολογισμό ενώ το Προεδρείο λέει, λένε οι Σοσιαλιστές. Όσον αφορά τώρα τις συνεισφορές, μονάχα από το ΕΛΚ αναφέρονται βάσει του άρθρου 7. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σα απολύτω και με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις προτάσεις όσον αφορά τα σημεία αυτά, έτσι ώστε καλύτερα να καταλάβουμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι μελλοντικέ συζητήσει και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, σε μια καλή συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη γιατί η φωνή μου δεν είναι και πάρα πολύ καλή σήμερα, λέει ο Μιλήτρια. Πρόεδρος, ε, ναι, υπάρχουν πολλές ε, πολλέ προτάσει. Βεβαίω εμεί εμείς, συγγνώμη, θα πρέπει να φτάσουμε με μια συγκεκριμένη θέση ε, αν είναι δυνατόν και βεβαίως θα πρέπει να το κάνουμε βάσει δημοκρατικής διαδικασίας. Γι' αυτό καλό είναι ε, να εκφραστούν οι πολιτικοί, να εκφραστούν ε, οι κοινοβουλευτικοί και οι βουλευτές αλλά οι αρμόδιες επιτροπές είναι αυτές οι οποίες θα αποφασίσουν μέσω της ψηφοφορίας και νομίζω ότι ο κατάλογος της ψηφοφορίας θα πρέπει μέχρι το Σάββατο το πρωί στην Ρώμη να ε, είναι ε, τέλειοι έτσι ώστε στη Ρώμη να υποβάλουμε συγκεκριμένο κείμενο. Ποιος θέλει να μιλήσει παρακαλώ κύριε Φέσσα. Θα μιλήσω στα γαλλικά γιατί έχω τις τροπολογίες στα γαλλικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τιτσιάνα Μπεγκίνε η οποία έκανε κατά την άποψή μου εξαιρετική εργασία, δύσκολη μάλιστα και περίπλοκη. Είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ Ευρωπα... Ε, Ευρωπαίων βουλευτών. Ε, να πω λοιπόν ότι πρόκειται για τροπολογίε οι οποίε προσπαθούν να βελτιώσουν το υφιστάμενο κείμενο. Αλλά για να είμαι απολύτω ε, ειλικρινή, πρέπει να έχουμε και ένα plan B μίλησα και με την Ινέσα Γιάλα και μου είπε και αυτή δεν θα προχωρήσει το πράγμα εάν ε, έχουμε διαφορετική θέση ανάμεσα σε Ευρωπαίους βουλευτές και εθνικούς ε, βουλευτές. Αυτή είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση ε, και επομένως δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε τα πάντα τώρα. Νομίζω ότι αν δεν λειτουργήσουμε σωστά δεν θα λειτουργήσει και η συνέλευση σωστά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, με τις τροπολογίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε κάπως να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ας πούμε, εμείς λέμε ε, να τελειώνει τέλη Ιουνίου ε, το οικονομικό έτος γιατί έχουμε ολομέλεια το Μάιο, τον Ιούνιο. Για να εγκριθεί λοιπόν ε, ο προϋπολογισμός είναι καλύτερος ο συντονισμός ε, ε, της Γενικής Συνέλευσης με την έγκριση του προϋπολογισμού. Αλλά αυτό είναι τεχνικό σημείο, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όσον αφορά τον κανονισμό τώρα της συνέλευσης. Νομίζω ότι η κεντρική ιδέα είναι ότι οι αντιπρόεδροι των επιτροπών ε, να μπορούν να συμμετέχουν στο διευρυμένο προεδρείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει η περίπτωση πολλών αντιπροέδρων από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά οι πρόεδροι είναι από τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε. Δεν είμαστε στο προεδρείο είναι σημαντικό λοιπόν το διευρυμένο Προεδρείο, ε, στο διευρυμένο να συμμετέχουν οι αντιπρόεδροι που συνήθως προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα, για να καθοριστούν οι συνεδριάσεις των επιτροπών θα πρέπει να υπάρχει η συμφωνία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Γιατί διαφορετικά αυτό που συμβαίνει είναι ε, ότι πολλές φορές ε, ε, συνεδριάζουν οι επιτροπές ας πούμε και συμπίπτουν οι συνεδριάσεις με την Ολομέλεια του Στρασβούργου και εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Θα πρέπει οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι να συζητούν από κοινού έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να επηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ημερομηνίε. Και αυτό είναι τεχνικής φύσεως το θέμα πάντως. Όσον αφορά τα οικονομικά, Στο, σχέδιο, στο προσχέδιο λέγαμε ότι η Επιτροπή Ad Hoc για τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού ε, που θα εγκρίνει ε, τον κανονισμό αλλά εάν είναι επιτροπή ad hoc και όχι μόνιμη ε, κάποια στιγμή θα πάυσει η λειτουργία της. Ε, εγώ πιστεύω ότι εμείς προτείνουμε το διευρυμένο προεδρείο και όχι το προεδρείο γιατί είπαμε ότι ως διευρυμένο προεδρείο έχουμε και εμείς παρουσία και το λόγο μας γιατί εάν πούμε ότι μόνο το προεδρείο θα πρέπει να αποφασίσει τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην εκπροσωπείται. Ε, και δεν είναι δυνατόν αυτό σε ένα σημαντικό θέμα και εν πάση περιπτώσει να μην το κάνουμε και τρομερό ζήτημα, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν καλύτερα να έχουμε και εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Καλό θα ήταν ίσως να συναντηθούμε με την Τιτσιάνα ε, και με τον υπεύθυνο από βουλευτή από πλευράς ε, της σοσιαλιστικής ε, ομάδας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι τόσο τρομερό το σημαντικό. Είναι τελικά να έχουμε κάτι λογικό και συνεκτικό και στο σύνολό του πιο εύκολο και πιο πρακτικό. Δεν έχουμε εδώ ιδεολογική και προσκόμματα. Ευχαριστώ πολύ. κινηθή σας. Ζητήσατε το λόγο. Ε, ναι, και άλλοι. Κάποιος άλλος ζητά το λόγο. Η κυρία Ροδρίγες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε πριν. Θα πρέπει να κάνουμε μία συνάντηση σε περιορισμένο κύκλο για να, συνα... για να συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα αποφα... και τι θα αποφασίσουμε. Αυτό που με ενδιαφέρει ωστόσο να σας ζητήσω είναι να προβλέψετε πορτογαλική μετάφραση την επόμενη φορά, διότι έχω συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις Ευρωμέντ και ποτέ δεν είχα μετάφραση στα πορτογαλικά. Πρόεδρος, ε, ναι, θα προωθήσουμε το αίτημά σας και θα δούμε αν από οργανωτική πλευρά αυτό είναι δυνατόν. Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για να κάνω μία πρόταση συγκεκριμένη. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε η Σέλφος Μπεγκίν, την οποία ευχαριστώ, γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές ε, ε, της αντιπροσωπεύσης του Κοινοβουλίου εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε και παλαιές εμπειρίες που θα μας ε, οδηγήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ απλώς να προωθήσουμε τα μέτρα τα οποία θέλουμε όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πράγματι αυτό που ακούστηκε προηγουμένως για το θέμα των αντιπροέδρων ε, είναι ε, σημαντικό όχι για να καπελώσουν ε, την συνέλευση οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά είναι καλό να γίνεται καλύτερη συζήτηση, να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε με κάποιο κοινά αποδεκτό κείμενο στην Ρώμη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περνιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια θα πω μόνο, πολύ γρήγορα. Και ευχαριστώ βεβαίω εξ αρχή την κυρία Μπεγκίν ε, για την προσπάθειά τη. Συμφωνούμε, όπως είπε και ο κύριος Πίσα πριν λίγο, ε, να κάνουμε κάποιες ε, προσαρμογές οι οποίες δεν είναι και ουσιώδεις, γιατί ήδη λειτουργεί το σύστημα αρκετά καλά όπως είπε και η κυρία Μπεγγίνε, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα, αλλά να διευρύνουμε κάποιες ε, αρμοδιότητες. Ε, έχω υποβάλει λοιπόν δύο προτάσεις ε, εντός των τρόπο λογιών. Το Περιφερειακό Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ενδυναμώσει την παρουσία του όσον αφορά κοινέ προβληματικές όπως είναι η ενεργεία, όπως είναι οι νέοι και ε, μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να καλούνται συστηματικά. Ε, νομίζω ότι και η Φιδερίκα Μογκερίνη θα πρέπει να έρχεται ε, στην αντιπροσωπεία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε μαζί να μπορούμε να καθορίσουμε ένα κοινό αφήγημα. Στις προτάσεις μας επίσης νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι επιτόπου αποστολές, ε, με κοινέ αποστολές βορρά-νότου, ε, με συγκεκριμένη θεματική, ε, στα πλαίσια των οποίων θα μπορούμε να διαπιστώνουμε και την πρόοδο διαφόρων έργων, αλλά και, την, και τον συντονισμό λόγων και έργων που δεν είναι προφανή πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Περνιό. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ακούσαμε την κυρία Μπεγκίν, ακούσαμε και τις παρατηρήσεις και επομένως εγώ θα πρέπει να σας δώσω ένα τρόπο ε, τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε μέχρι να φτάσουμε στην, στην Ολομέλεια της ε, Ρώμης. Ε, έχουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα κείμενο το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της μεγαλύτερης δυνατής συνένεσης. Σάββατο πρωί νομίζω στην Ολομέλεια θα πρέπει να έχουμε ήδη μια πρόταση η οποία θα, συγκεκριμένη η οποία θα υποβληθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ορίσουμε προθεσμία συγκεκριμένη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε το υπόλοιπο τούτης της εβδομάδας και την επόμενη εβδομάδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς προτάσεις, ε, αν όχι θα υποβάλω εγώ μία πρόταση. Κυρία Μπεγκίν, θέλετε να προτείνετε κάτι. Eh, έχουμε τις εξής ε, δυνατότητες. να πούμε εξ αρχής ε, ότι μπορεί να γίνει μια τεχνική προπαρασκευαστική εργασία από τους ε, υπαλλήλους και την επόμενη εβδομάδα, τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας έτσι ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο, να προσπαθήσουμε ε, να κάνουμε μια τεχνική συνάντηση με εκπρόσωπο από κάθε ομάδα έτσι ώστε και οι ε, πολιτικές ομάδες ε, να κάνουν τις εσωτερικές τους συζητήσεις και να στείλουν έναν εκπρόσωπο στη μήνυ ομάδα εργασίας. Κύριε. Συμφωνώ απολύτως με αυτό, λέει ο κύριος Φίσας. Με τον τρόπο αυτό οι υπάλληλοι μπορούν λίγο να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να προχωρήσουμε ε, ε εγώ ε, ε, υπέβαλα την ε, τροπολογία για την μετατόπιση της συνέλευσης γιατί θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου πρώτα θα έχουμε την συνέλευση και μετά θα έχουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και εξ ανάγκης θα έχουμε πλέον ένα προσχέδιο προϋπολογισμού γιατί δεν θα μπορεί να γίνει ε, η έγκρισή του κανονικά από την Γενική Συνέλευση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείναμε ε, να αλλάξει η ημερομηνία της ε, συνέλευσης έτσι ώστε ο γενικός προϋπολογισμός να εγκρίνεται τελειωτικά από την Ολομέλεια. Κύριε Φίσα, νομίζω ότι, Φίσας, νομίζω ότι λέει ο Πρόεδρος δεν θα είναι δύσκολο να βρεθεί μια τεχνική λύση ε, ε, βάσει αρχών ε, λογικής απλής. Έτσι. Θα, θα, βρεθεί μια κοινή θέση. Κύριε Πυρνιό ως συντονιστής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Μπεγκίν. Λοιπόν, εγώ λέω να προχωρήσουμε ως εξής, λέει ο Πρόεδρος. Να ζητήσουμε από την Γραμματεία να ε, κάνει, ε, να, ε, ένα τεύχος με όλες τις τροπολογίες και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων ε, και της Προέδρου Μπεγκίν ε, και της ε, Γραμματείας έτσι ώστε να βρεθεί ένα κείμενο γιατί άλλωστε και η Γραμματεία θα χρειαστεί και κάποιες μέρες έτσι ώστε το Σάββατο να καταφέρει να έχει Σάββατο πρωί να έχει ένα κείμενο. κοιτάξτε, εμείς έχουμε και ένα προηγούμενο που είναι η ομάδα εργασίας της Παρασκευής αυτό είναι το Προεδρείο, λέει ο Προεδρο. Όχι, όχι, το πρωί έχουμε και ομάδα εργασία μαζί με, τις, ε, με τα άλλα κοινοβούλια. Γιατί τη μεταρρύθμιση δεν την προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρασκευή, λέει ο Πρόεδρο. Ναι, αλλά από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή νομίζω ότι μπορούμε. Αλλιώ, ε, εάν θεωρείτε ότι δεν τα καταφέρνουμε, Τρίτη να γίνει καλύτερη συνεδρίαση. Τρίτη. Ναι, και, το, και η Γραμματεία επιβεβαιώνει ότι είναι καλύτερα την Τρίτη. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ήδη από τώρα ότι την Τρίτη θα έχουμε τη συνάντηση με, ανάμεσα στην Πρόεδρο Μπεγίν, ε, τους ε, ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, τους βουλευτές που θέλουν να συμμετάσχουν και τη Γραμματεία έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε μία συμβιβαστική λύση. Από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή θα επεξεργαστούμε το κείμενο το οποίο θα επιβληθεί στην ομάδα εργασίας της Παρασκευής. Συμφωνείτε? Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε? Όχι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Νομίζω ότι αυτή η συνεδρίαση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μπεγκίνε και το λέω βλέποντας την κατάσταση απ' έξω, ε, δεν αφορούν ε, σημαντικά ιδεολογικά ζητήματα, αφορούν πρακτικά απτά θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν βάσει της λογικής. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι δύσκολο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις... Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.